Άρχισαν οι ψηφοφορίες. Θα περάσουμε τώρα. Στις επεξηγήσεις ψήφου. Ce ne sono 23.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari che... Λοιπόν, οι βουλευτές οι οποίοι θέλουν να ανακοινώσουν, να, που δεν θέλουν να κάνουν ανακοινώσεις και επεξηγήσεις, παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα. Ξεκινάμε με την έκθεση Αουστρεβίτσιους. Μάνικινς για ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Μαμίκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, εμείς υποστηρίζουμε το ψήφισμα για τη Μολδαβία και εγώ το υπερψήφισα και νομίζω είναι σημαντικό για το λαό της Μολδαβίας όχι μόνο ε, γιατί θα έχει και την ευκαιρία κάποια στιγμή να προσχωρήσει στην Ένωση Μολδαβία, αλλά ε, διότι αυτό είναι και κίνητρο και ενθάρρυνση για να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Οι πολιτικοί δεν μπορούν πάντα να επιβάλλουν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά τώρα έχουν περισσότερα επιχειρήματα. Γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να, εργαστεί στη, να δουλέψει στην πράξη. Πριν από 15 χρόνια θυμάμαι τη Λετωνία, τη χώρα μου. Στην πορεία της στην προεταξιακή έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά, αλλά προσεκτικά ο κόσμος περιμένει πάντα αποτελέσματα. Και βάσει αυτών μας κρίνει. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τη Μολδαβία και να ε, ξεκινήσει ένας διάλογος με την ε, υπερδνηστερία μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, η βία δεν είναι λύση. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι και εισηγητής, ξέρετε, για τη Γεωργία ε, και υποστηρίζω ε, αυτές τις εργασίες και σας παρακαλώ ε, στην επόμενη Ολομέλεια να υποστηρίξετε και τη δική μου έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ όσοι δεν θέλετε να κάνετε επεξηγήσεις ψήφου να αποσυρθείτε ησύχως. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Αλλά παρόλα το λόγο έχει ο κύριος Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χάρηκα πολύ που μπόρεσα να στηρίξω σήμερα στην ψηφοφορία τη Συμφωνία Σύνδεσης με τη Μολδαβία. Εγώ είμαι Τσέχος και θυμάμαι ακόμη πόσο υποφέραμε ε, τώρα θα ενδυναμωθούν οι εμπορικές σχέσεις και θα βελτιωθεί το πολιτικό πλαίσιο. Η Μολδαβία είναι τώρα στο δρόμο προς την Ένωση και μπορεί να προσβλέπει σε αυτήν. Δεν χρειάζεται να εξαρτάται από τη Ρωσία. Αλλά νομίζω ότι στο μέλλον πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Εγώ ήμουν υπουργό δικαιοσύνης στην Τσεχία και είχα τη χαρά να διαπραγματευθώ με τους ε, Μολδαβούς για την μεταρρύθμιση του δικαστικού των συστήματος για την εφαρμογή του κράτους δικαίου, σωστών δομών κλπ. Και γι' αυτό συγχαίρω τη Μολδαβία για την σημερινή ψηφοφορία. Ο κύριος Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ με μεγάλη χαρά ε, ψήφισα και υποστήριξα τη Συμφωνία Σύνδεσης. Εγώ είμαι από τη Σλοβενία. Όπως και άλλοι συνάδελφοι θυμάμαι εκείνες τις εποχές ε, στην προεταξιακή πορεία προς την Ένωση. Ε, συμφωνώ και με το ελεύθερο εμπόριο και το υποστηρίζω για τα όπορο κυπευτικά. Αυτά είναι θέματα της Επιτροπής Γεωργίας. Και ε, πρέπει να σας πω ότι και εγώ αγρότης είμαι. Και μάλιστα έχω τέτοιες καλλιέργειες ε, οποροκυπευτικών, αλλά θα υποστηρίξω τη συμφωνία. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι το ελεύθερο εμπόριο για τον κόσμο, για τους ανθρώπους επιτόπου και είναι και ένα θέμα τιμής. Και σε αυτό το σημείο για την ε, Δημοκρατία της Μολδαβίας δεν συζητήσαμε το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα κάνει απικία της στη Μολδαβία, η Ρωσία θα κάνει απικία της στη Μολδαβία για την καλύτερη ζωή των ανθρώπων ενδιαφερόμαστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίριο δεν είναι εδώ. Περνάμε στον κύριο Χάναν για ένα λεπτό. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Κάθε χώρα που γυτνιάζει με τη Ρωσία έχει αισθανθεί την πίεση που της θέτει ο Πούτιν καμιά φορά με βάση το πετρέλαιο και το αέριο, άλλες φορές όπως στην Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Βεσαραβία, με τη μορφή στρατιωτικής κατοχής. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκε η Δύση σε όλα αυτά και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δυστυχώς μια δίθεν μετριοπάθεια και μέση οδός ο Πούτιν θέλει να δημιουργήσει μια Ευρω... ευρωασιατική ένωση ελευθέρων συναλλαγών από τη Λισαβόνα μέχρι τα Ουράλια. Όλα αυτά βέβαια χωρίς κανένα σχέδιο αντιμετώπισης από μας και αυτά τα πληρώνουν οι λαοί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως εγώ δεν ψήφισα υπέρ της συμφωνίας ε, σύνδεσης, αλίμονο. Δεν πρόκειται να ψηφίσω ε, για μια νέα απικία ε, των πολυεθνικών εταιριών που ανοίγουν νέες αγορές. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Ο συνάδελφος Τόκιος που είναι από την Τρανσιλβανία, Ούγγρος, είναι υπέρ γιατί ε, θεωρεί ότι είναι λύση για την Ενωμένη Ευρώπη και η Ενωμένη Ευρώπη είναι λύση για τις κοινότητες. Δεν μπορούσα να κάνω ερώτηση με μπλε κάρτα γιατί δεν μου δώσατε το λόγο. Τώρα μπορώ να του πω και σε όλους ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει, δεν είναι λύση αυτή η συμφωνία. Διότι αν ήταν τέτοια λύση θα είχαμε αυτονομία ε, στις περιφέρειες και αυτοδιάθεση και της ε, Τρανσιλβανίας. Η Ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Ούτε τα διατάγματα Μπενές ε, στην Τσεχία και την Τσεχοσλοβακία γενικότερα δεν λύθηκε αυτό. Ούτε στις διαπραγματεύσεις με τη Σερβία κάναμε τίποτα για την αυτοδιάθεση της Βοηβοδίνας και όταν μιλάμε για την Ουκρανία ποτέ δεν αναφερόμαστε στην αυτοδιάθεση των ε, Ούγγρων που ζουν στη Δυτική Ουκρανία. Mr. Chairman, our party and our group have opposed. Εμείς σαν κόμμα και σαν πολιτική ομάδα ήμασταν κατά της τροπολογίας και την πορεία της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκαθαρίσαμε ότι για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σαν ένας επιθετικός απεικιοκράτης. Όπως οι χώρες σαν τη δική μου που στο παρελθόν είχαν αποφασίσει να ελέγχουν οικονομικά χώρες στη σφαίρα επιρροής τους. Το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγχει τη Μολδαβία. Κάνοντας το αυτό συμπεριφέρεται με παιδικό τρόπο λέγοντας ότι θα φοβήσουν τη ρωσική αρκούδα που και αυτή έχει μια ζώνη επιρροή στην περιοχή. Αντί να είναι λογική και διαπραγματευτική απέναντι στη Ρωσία, ε, νομίζουν ότι επιτιθέμενοι στη Ρωσία με τον τρόπο αυτό ε, θα εκδικηθούν για αυτά που έκανε η Ρωσία στο παρελθόν. Αυτό δεν έχει λογική σαν διπλωματική ενέργεια ούτε σαν πολιτική ενέργεια. Περνάμε τώρα στην σύσταση για την σύσταση για τη Μολδαβία. Ο κύριος Χάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, δεν θέλει τον λόγο. Γκίλ. Ευχαριστώ. Μια συμφωνία σύνδεσης είναι ένα βήμα πέραν από την πλήρη ένταξη. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μολδαβία ως προς τις σχέσεις της με τη Ρωσία και την Ένωση για να μην αναφερθώ καθόλου για, στην ανθρωπιστική κρίση που βλέπουμε στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλα τα συμβαλόμενα μέρη να κρατήσουν λογική στάση. Η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Μολδαβία ιδιαίτερα ως προς την ιστερία, μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο την κρίση και σκεπτόμενοι αυτό καταψηφίσαμε. La parola Frunzulica per un minuto. Κύριος Φρονζουλίκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα πάρα πολύ τη Συμφωνία Σύνθεσης Ένωσης και Μολδαβίας διότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό βήμα στον δρόμο για την επανένταξη εγώ θα έλεγα της Μολδαβίας στην Ευρώπη γεωγραφικά και πολιτιστικά ήταν αναπόσπαστο τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πολιτικά και γεωστρατηγικά επανέρχεται τώρα στην Ευρώπη όπου ανήκουν οι άνθρωποι της και οι πολίτες της και θα επωφεληθούν πάρα πολύ από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας χρειάζονται και αξίζουν την υποστήριξή μας. Περνάμε τώρα στην ειρηνευτική διαδικασία στην Βόρεια Ευλανδία Άντερσον. Το λόγο έχει ο επόμενος. Κάθε. Uh, um, I voted in favor of... Εγώ ψήφισα υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας, του ψηφίσματος για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία και θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για την έγκρισή του με τέτοια συντριπτική πλειοψηφία. Προέρχομαι από μια πόλη στα νότια σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας προς τα σύνορα με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Ξέρω ότι πόσο αρνητική είναι η διαίρεση της χώρας και η σύγκρουση καθώς και η απώλεια τόσων πολλών ζωών λόγω της σύγκρουσης αυτής. Επίσης όμως γνωρίζω τις δυσκολίες που έχουμε διότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φορολογικά καθεστώτα, δύο νομίσματα, δύο υγειονομικά συστήματα και θα ζητούσα από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας στηρίξουν για να μπορέσει η οικονομία του συνόλου της Ιρλανδίας να αναπτυχθεί και να συνεχιστεί η επιτυχής ειρηνευτική διαδικασία. Μπόιλαντ. Μπόιλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του σε αυτό το ψήφισμα ψήφισα υπέρ και νομίζω ότι η στήριξη που φάνηκε σήμερα δείχνει ότι υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον και υποστήριξη για τον τερματισμό των παρελθόντος. Ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης Χάρηκα ιδιαίτερα που έγινε λόγος για την ανάγκη περισσότερης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για να γίνει βιώσιμη η ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι η κυβέρνηση των συντηρητικών προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει περικοπές στα επιδόματα για τους φτωχότερους. Εμείς με ολόκληρη την εργατική τάξη στον βορρά της Ιρλανδίας αντιτιθέμεθα στις περικοπές αυτές. Και γι' αυτό ζητώ από όλα τα κόμματα στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας να πράξουν το ίδιο. Κύριε Χάρα, ευχαριστώ. Πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος Σούλτς είπε ότι ήταν μεγάλο κατόρθωμα η ειρηνευτική αυτή διαδικασία. Βεβαίως είναι κατόρθωμα. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε να επιστρέ... θέλει κανείς να επιστρέψει στη βία που κατέστρεψε τη ζωή μιας ολόκληρης γενιάς. Και εγώ έχω τέτοια ενδιαφέροντα γιατί η οικογένειά μου είναι η μισή καθολική και η άλλη πρεσβυτεριανή. Δεν πρέπει όμως τα κόμματα που είναι στην εξουσία να εφαρμόζουν πάντα τη συνταγή των δημοσίων θέσεων και των δημοσίων δαπανών παραπάνω και από τη Σοβιετική Ένωση. Όλοι ξέρουμε, επειδή είμαστε δημοκρατικοί πολιτικοί, ότι η αντιπολίτευση είναι κάτι που μαστιγώνει τη δημοκρατία και την προωθεί, γιατί έχει τα αντισχέδια. Χωρίς αντιπολίτευση δεν υπάρχει δημοκρατική κοινωνία. Ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ενευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι κάτι ε, το υποδειγματικό αν σκεφτούμε τις καταστάσεις του παρελθόντος. Θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ε, υποδειγματική στάση τα δύο μέρη και αυτό θα εμπνεύσει και άλλες κοινότητες ως διαδικασία ειρήνευσης η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία αλλά και στην πρόληψη των συγκρούσεων ιδιαίτερα. Και στα κράτη-μέλη της Ένωσης και στα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν πολλά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με ε, τις κακές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων που δεν έχουν ε, ρυθμιστεί και διευθετηθεί. Θα πρωταγωνιστήσουμε εμείς ε, για να υπάρξει μια σταθερή κοινωνία και στη Βόρεια Ιρλανδία και μπορεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί διάφορες ε, διακοινωτικές διαφορές ε, και στις υποψήφιες χώρες αλλά και στα κράτη-μέλη της ίδιας της Ένωσης και πρέπει να παίξει, ε, είπαμε, πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Ο κύριος Σιτουργάηθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η Ισπανική Αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος καταψήφισε την έκθεση για τη Βόρεια Ιρλανδία για διάφορους λόγους. Θεωρούμε ότι η απουσία από την έκθεση αναφοράς στα θύματα της τρομοκρατίας και η απόρριψη της προφορικής τροπολογίας ε, που θα ανέφερε ρητά αυτό για να μην υπάρξει ατιμορρησία είναι αρκετοί λόγοι για να καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Επιπλέον όμως θέλω να θυμίσω κύριε Πρόεδρε ότι έγιναν σχόλια χτες ε, το βράδυ στη συζήτηση που ε, συνέκριναν τη Βόρεια Ιρλανδία με τη χώρα των Βάσκων. Θέλω να θυμίσω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία υπήρξε ένοπλη σύραξη μεταξύ δύο μερών. Στην χώρα των Βάσκων Μόνο υπήρξε και υπάρχει ένοπλη σύραξη από μία πλευρά που είναι οι δολοφόνοι τρομοκράτες της ΣΕΤΑ που έχουν ε, σκοτώσει εκατοντάδες αθώα θύματα. Και δυστυχώς αυτή η τρομοκρατική συμμορία όπως όλοι γνωρίζουμε συνεχίζει τη δράση της. Δεν θέλει να εγκαταλείψει τα όπλα ούτε να τα καταθέσει ούτε ε, να ε, διευκολύνει την εξυχνίαση πάνω από 300 δολοφονιών που έχουν μείνει εγκλήματα χωρίς τιμωρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Mr. Kelly, you have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της χθεσινής συζήτησης και για την ψηφοφορία σήμερα και φυσικά υποστηρίζω τις προτάσεις αυτές. Εκτιμώ το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και να σημειώσω εδώ ότι έχουν ήδη επιτυλιστεί σημαντικά βήματα προόδου. Ελπίζω η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί στο μέλλον. Σχετικά με τις προφορικές τοπολογίες, κατανοώ αυτό το οποίο ε, ε, εννοήσατε πριν από τις τροπολογίες. Είχαμε πει όμως ότι εμείς δεν θα ε, είχαμε συνεννοηθεί ότι δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε περαιτέρω τέτοιες προτάσεις γιατί είναι κάτι το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά την Βόρεια Ιρλανδία. Ναρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι Βάσκος και ο πατέρας μου ζούσε στην ε, χώρα των Βάσκων και τον απείλησαν ότι θα το σκοτώσουν γιατί δεν πλήρωσε το εκβιαστικό τίμημα της ε, τρομοκρατικής συμμορίας. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ παραλληλισμό και σύγκριση με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να λυθούν άλλες συγκρούσεις. Πρώτον, ήταν ε, αντιδημοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το ψηφισμό. Ούτε τροπολογία δεν μας αφήνανε να κάνουμε. Αν ε, είχε ε, γίνει δεκτή ε, η ε, τροπολογία της συναδέλφου της οποίας σκότωσαν τον αδελφό λόγω αυτής της σύγκρουσης εμείς θα είχαμε ε, συμφωνήσει. Τρία πράγματα. Πρώτον, δεν γίνεται λόγος για τα θύματα βάζουμε στην ίδια μοίρα ε, θύτες και θύματα, δολοφόνους και δολοφονηθέντες και υπάρχει ατιμορρησία. Η παράγραφο Δέλτα που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση ε, και αμοιβαία ε, σεβασμός και τα λοιπά μεταξύ δολοφόνων και δολοφονηθέντων καμία. Γιατί στη χώρα των Βάσκων δεν είναι διακοινωτική σύραξη αλλά ήταν κάποιοι που είχαν άλλα μυαλά από του τρομοκράτε και του σκότωσαν. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος για τις ενέργειες ε, της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Μπόγκοβιτς. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα πράγματι συζητήσαμε στην συνάντηση με την διακοινοβουλευτική με την Τουρκία μιλήσαμε για την Τουρκία και για τον δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο μας αποσχόλησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της ε, εβδομάδας. Μιλήσαμε για τις ε, σχέσεις της ειρηνικές ανάμεσα στην Κύπρο και την Τουρκία και στην βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα της της Κύπρου. Πρέπει λοιπόν να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε και τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός του Κυπριακού όπως το θέμα το Συριακό σαν παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Στις αρχές του 90 οι δύο πλευρές στην Κύπρο πλησίαζαν σε λύση. Δηλαδή αντάλλαγμα γη για ειρήνη. Θα παρέδιναν μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα οι Τούρκοι για να διατηρηθεί η ειρήνη. Και καθώς επρόκειτο να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Η Ένωση αναγνώρισε μονόπλευρα τη μία πλευρά και αμέσως η άλλη έχασε κάθε θέληση να διαπραγματευτεί και χάθηκε η ευκαιρία. Δεν έφταιγε η Τουρκία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση με την μονομερή της αντιμετώπιση. Μία από τις δύο κοινότητες υπερψήφισε το σχέδιο ειρήνευσης τιμωρήθηκε και η άλλη το αρνήθηκε και επιβραβεύτηκε. Εδώ υπάρχει μια βασική αδικία και προς την Τουρκία που είναι φίλος και σύμμαχός μας και τήρησε τέτοια αμυντική στάση κατά των Μπολσεβίκων και του Μπολσεβικισμού. Δεν είναι τρόπος αυτός να φέρεται κανείς τους συμμάχους του. Mr. Ζαχραντήλ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εγώ λυπούμαι ε, που ενέκρινε σήμερα το ΕΛΚ τη συγκεκριμένη έκθεση. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, είναι μονομερές, ε, μεροληπτικό και δεν θα βοηθήσει θετικά να λυθεί αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Και μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που θα σταματήσει η Τουρκία κάθε προσπάθεια για διμερείς συνομιλίες. Ως πρόεδρος και ε, του κόμματός μας που είναι μέλος και το μεγαλύτερο κόμμα της Τουρκίας το ΑΚΠ πρέπει να σας πω ότι καταψήφισα την έκθεση αυτή γιατί δεν συμφωνώ καθόλου. Ευχαριστώ. Πρόταση ψηφίσματος για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Άναν πάλι. δημιουργούνται συνεχώς όλο και καινούριε χώρες. Σπάνε οι παραδοσιακές αυτοκρατορίες και έχουμε νέα ανεξάρτητα κράτη. παντού, εκτός από την Ήπειρο αυτή, όπου εδώ τα πράγματα πηγαίνουν προς την ανάποδη πορεία θα έλεγα και γίνονται όλο ένα και πιο συγκεντρωτικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις μιας μικρής ελίτ. Ζούμε στη μόνη ε, περιοχή του πλανήτη η οποία δεν έχει καμία ε, ένδειξη οικονομικής ανάκαμψης. Ε, τα προβλήματα της Ευρώπης είναι γνωστά ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη και βλέπουμε ότι δεν θα βγουν εύκολα μετά από τόσα χρόνια στασιμότητας από την κατάσταση αυτή γιατί αντικαταστήσαμε τα κράτη από συγκεντρωτικά συστήματα. Είμαστε το μόνο μέρος του κόσμου το οποίο βυθίζεται. Τζουφρίντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εκ νέου ότι υπερψήφισα την έκθεση όπως είπα και χθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Νότιο Σουδάν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν έχουν σταματήσει οι μάχες και υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που μας λέγουν ότι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κάτοικοι της περιοχής θα φυγούν ε, ιδιαίτερα μετά από, την, ε, ε, μετά από τη νέα περίοδο βροχών που θα ξεκινήσει στην περιοχή και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται σε πρόχειρα καταλήματα στην Αιθιοπία κυρίως θα αντιμετωπίσουν τρομερά προβλήματα αν και βοηθά το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς έτσι ώστε να συνεχίσουν και τα Ηνωμένα Έθνη να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την επίλυση μιας δύσκολης κατάστασης. Ευχαριστώ η κυρία Κιέντζε. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Κιέντζε. Κύριε Πρόεδρε, με το ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει μια νέα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση στη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν μια περιοχή μαρτυρική, δύο δεκαετίες συγκρούσεων εκατομμύρια νεκρών. Από το 2011 υπήρξε ελπίδα για το λαό της ε, περιοχής του Νοτίου Σουδάν, αλλά υπάρχουν προβλήματα και υπήρχαν από τότε οι σπόροι ανθρωπιστικής καταστροφής. Χιλιάδες παιδιά δεν μπορούν να πηγαίνουν σχολείο, τα προβλήματα διατροφής είναι τεράστια, υπάρχουν προβλήματα με τους πρόσφυγες γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να αναγκάσει όλους τους εμπλεκομένους να θέσουν τέλος στην σύραξη η οποία υπονομεύει το σύνολο της περιοχής και τις γειτονικές χώρες. Είναι απαραίτητο επίσης και η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα οι γυναίκες, πρέπει να πάρουν μέρος στις ειρηνευτικές διαδικασίες, όπως επίσης και να συζητήσουμε για το τι θα γίνει μετά το τέλος των σειράξεων σχετικά με την ανικοδόμηση της χώρας. Δυστυχώς τα όπλα εξακολουθούν ε, να ρέουν στην περιοχή και η κατάσταση χειροτερεύει. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν να προσυπογράψει τη σύμβαση του Κοτονού στα πλαίσια της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Ευχαριστώ κυρία Κιέντζε. Ο κύριος Κέλλη, είστε ο τελευταίος ομιλητής για σήμερα. Ναι, αλλά και ο καλύτερος ίσως. Λοιπόν, όπως και οι προλαλήσαντες θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε ως πρόεδρος της σημερινής συζήτηση. Επίσης, χάρηκα ιδιαίτερα που μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή και νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Κοινοβούλιο για να χορηγήσουμε ως το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη στο λαό του Νότιου Σουδάν. Όταν αποσχίστηκε η περιοχή αυτή πριν από τρία χρόνια, νόμιζε οι κάτοικοί ότι θα έχουν λαμπρό μέλλον. Άλλοι όμως ανησυχούσαν ιδιαίτερα γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το νέο αυτό κράτος εύκολα και αυτό έγινε. Γι' αυτό ζητούμε από τις αρχές του Νότιου Σουδάν να λύσουν τα προβλήματά τους και να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσα διαθέτουν για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους. Με μεγάλη χαρά λοιπόν έδωσα την υποστήριξή μου και σας ευχαριστώ ξανά για τη δουλειά που κάνετε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Εφόσον δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, τα ψηφίσματα τα οποία, τα ψηφίσματα τα οποία έγιναν δεκτά θα αποστελούν ε, εκεί που χρειάζεται και τέλος της σημερινής συνεδρίασης.